Notre Αρχίζει η συνεδρίαση και αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση θεωρώ ότι η μερίσια διάταξη όπως σας έχει προταθεί υιοθετείται και θα ήθελα να σας ανακοινώσω τις αποφάσεις των ε, συντονιστών τις οποίες μόλις πήραμε Καταρχήν, μάθαμε ότι έγινε ένα έμβασμα για τη χρηματοδότηση της, ε, του θέματος των οδηγών της ε, ενσωμάτωσης των οδηγών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ξέρετε, η Ολομέλεια είχε ψηφίσει ένα αποθεματικό Προτείνω λοιπόν να προετοιμάσουμε μια επιστολή που θα υπογραφεί από κοινού με τον κύριο Ταρό για τον προϋπολογισμό του 17 και τον ΔΕΠΡΕ για τον προϋπολογισμό του 16 καθώς και από εμένα τον ίδιο και τώρα όσον αφορά τους διάφορους εισηγητές για τις εκθέσεις, τις γνωμοδοτήσεις και τις δικές μας πρωτοβουλίες όσον αφορά καταρχήν την προσαρμογή για τις ε, πλήρωμες για την κοινή αγροτική πολιτική προς τους γεωργούς, οι εισηγητές θεώρησαν ότι εδώ δεν υπάρχει λόγος να προετοιμάσουμε μια δική μας γνωμοδότηση. Όσον αφορά το Investing in Jobs and Growth, και την ε, μεγιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Συνοσφοράς καθώς και το άρθρο 16.3 του CPR θα υποβάλουμε γραμμοδότηση. Οι σοσιαλδημοκράτες είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν αυτή τη γνωμοδότηση. Το θέμα τώρα της, ε, του κανονισμού ο κύριος Γκάιερ θα αναλάβει την έκθεση αυτή ως εισηγητής. Τώρα, τις ε, κατεξοδότσι πράξεις. Ε, όσον αφορά την κάλυψη των εγγυήσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για δάνεια που θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς την Λευκορωσία, πρόκειται για μία απόφαση για την οποία θεωρούμε ότι πρέπει να υποβληθεί εδώ μία πρόταση, αλλά προηγουμένως θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση. Εάν αύριο, μετά το πέρας της συζήτησης, αποφασίσει η κυρία Κάρτες πάλι μόνιμη εισηγήτρια, ότι πρέπει να το αναλάβει η ίδια, θα το κάνει. Αλλιώς θα το αναλάβω εγώ σαν πρόεδρος. Τώρα, όσον αφορά την αναβολή της πρότασης σχεδίου προπολισμού για το 2017, διότι παραδοσιακά υποβάλλεται το Μάιο, όμως για να υπάρξει μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά τις πιστώσεις για τους πρόσφυγες, την υποδοχή των προσφύγων και το θέμα της ε, μετανάστευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η αξιολόγηση με όλες τις λεπτομέρειες δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του Ιουνίου. Οπότε το σχέδιο προπολογισμού για το 2017 θα μπορέσει να μας υποβληθεί τέλος Ιουνίου του 2017. Μπορείτε να σχολιάσετε όπως θέλετε αυτήν την αναβολή, προσωρινή αναβολή. Εν πάση θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο Κινδυνεύουμε βεβαίως να μην είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε και τον τριμερή διάλογο για τι 13 ε, Ιουλίου. Αυτό είχε αποφασιστεί το 2014 μετά το τέλος των ε, ευρωπαϊκών εκλογών. Ο ειδικός εισηγητής ε, στέλνει μια επιστολή στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και βεβαίως σε αυτό συνοδεύονται, με αυτό υποβάλλονται συγγνώμη και όλες οι γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορέσουμε βεβαίως να αναβάλουμε τον τριμερή διάλογο, να ορίσουμε μια νέα ε, ημερομηνία. Αυτό όμως ε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει πριν τις 22 Ιουλίου, η ημερομηνία κατά την οποία διακόπτονται οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα αυτό θα δικατασταθεί και από την ε, μεταγενέστερη απόφαση της εισηγήτρια του εισηγητή. Το θέμα τώρα της μεταναστευτικής κρίσης και των προσφύγων είχε προβλεφθεί στις 15 Ιουνίου η συζήτηση στην ε, ΑΦΕΤ. Αυτό θα γίνει στις 30 Ιουνίου, αναβάλλεται δηλαδή. Όσον αφορά το διαρθρωμένο διάλογο, τον ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε τον κατάλογο. Εδώ θα προσθέσουμε και το θέμα της ε, φορολογικής δυνατότητας της Ευρωζώνης. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να οργανωθεί ένα εργαστήριο, ένα workshop για την αναθεώρηση του οικονομικού κανονισμού. Και αυτό θα μπει στην ημερήσια διάταξη το συντομότερο δυνατόν, διότι όλοι συμφωνούμε, πιστεύω ότι χρειάζεται απλοποίηση αυτός ο κανονισμός έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού των διαδικασιών, μόνιμος εισηγητής για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όλων των ε, χρηματοπιστωτικών εργαλείων, η κυρία Γκάρτε Σαμπάλ, θα προχωρήσει με την προετοιμασία του θέματος αυτού. Αυτές είναι οι αποφάσεις των ε, συντονιστών. Νομίζω ότι έχουν ζητήσει πέντε λεπτά διάλειμμα οι σοσιαλιστές για να μοιράσουν τον κατάλογο ψηφοφορίας. Καλά κατάλαβα. Non. Cette demande n'est pas confirmée. Όχι. Bien, nous allons passer. Εντάξει. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Confirmé? Donc la séance est suspendue pour... Διακόπτουμε για 5 λεπτά και στις 4.30 θα ξαναρχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Προτού να περάσουμε στις ψηφοφορίες, θα ήθελα να διαβεβαιωθώ ότι τα πρακτικά της 4ης Απριλίου δεν ε, έχουν ε, παρατηρήσεις από πλευρά σας, ενστάσεις και μπορούν άρα να γίνουν δεκτά. Παρακαλώ να πάρετε τις κάρτες σας ε, για να τις βάλετε στα μηχανάκια ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε κατά πόσο λειτουργούν ορθά. Άρχεται η ψηφοφορία, δοκιμαστική, πέρας αυτής. Σας ευχαριστώ. Λειτουργεί το μηχάνημα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε επί της έκθεσης κυρίας Γιάτεν Μάκη. Τροπολογία υπερθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία υπερθμών 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπερθμών 3. Υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογή υπερθυμών 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή υπερθυμών 5 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογή υπερθυμών 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή Υπαριθμούν 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία υπαριθμών 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Υπαριθμόν 11. ψηφί Ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπαριθμόν 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπορή υπαριθμό 13. Ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Έγινε δεκτή. Υπαριθμό 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Υπαριθμό 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία υπαριθμό 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτεί Και τώρα επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία, το κείμενο εγκρίθηκε 22 ψήφοι υπέρ 4 κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα Περνάμε στην ψήφιση της έκθεσης ε, της κυρίας Νιριάντα, τροπολογή παριθμών 1, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογή υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογή υπαριθμών 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Υπάρχουν 4 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία υπάρχουν 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Υπάρχουν 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπάρχουν 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία υπαριθμών 9 υπέρ α συγγνώμη τροπολογία υπαριθμών 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές ε, θα επαληθεύσουμε άρχιτη ψηφοφορία Σκρουτάει κλού. Πέρα ψηφοφορίας απορρίφθηκε 13 με 12. Ήταν η τροπολογία 8, παίρναμε στην 9 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της 9 ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία υπαριθμών 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία υπαριθμών 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή, προπολογία υπέρ 13 υπέρ, κατά, θα επαληθεύσουμε. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται 14 ψήφι κατά 10 υπέρ. Ήταν η τροπολογία υπαριθμών 13. Τώρα υπαριθμών 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία υπαριθμών 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Υπερθμό 17. Υπέρ κατά αποχές δεκτή παίρνουν 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή υπέρθμον 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή υπέρθμον 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Επί του συνόλου με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Σκοτάει Έληξε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά. σε Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Στην εισηγητή, συγγνώμη. Και τώρα περνάμε στην έκθεση του κυρίου Ζων Πολ Ντενανό. Συμβαστική τροπολογία υπερθυμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, συμβαστική τροπολογία υπερψηφίστηκε, άρα η τροπολογία 1 καταπίπτει. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία υπερθυμών 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία το πρώτο τμήμα αυτής ψήφι υπέρ κατά θα ελέγξουμε άρχιτη ψηφοφορία Έλλη ψηφοφορία. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι τα σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα. Έλλειξη ψηφοφορία. Το δεύτερο τμήμα υπερψηφίστηκε. 20 προς 6. Τροπολογική υπαριθμών 5. σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αυτή ψήφι Κατά. Αποχές. Το πρώτο τμήμα απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα. Προπολογή υπέρ 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ. η τροπολογία 6 απορρίπτεται μόνο 7 τώρα ψήφι πέρ. κατά Αποχέ. απορρίπτεται η τροπολογία μόνο 8 ψήφι πέρ. κατά Αποχέ. εγκρίνεται υπαριθμόν 9 τροπολογία ψήφι υπέρ κατά Αποχέ εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Η συμβαστική τροπολογία 2 εγκρίνεται, ω εκ τούτου η 10 καταπίπτει. Η τροπολογία 11 υπέρ. <clears throat> κατά. Αποχές. Κάποιοι δεν ψήφισαν, δεν ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε επί της 11 ηλεκτρονικός άρχη ψηφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε 17 ψήφι πέρ, 8 κατά. Παρακαλώ να γύρετε τα χέρια σας. Το που 12 υπέρ. Κατά. Αποχέσω. Εγκρίθηκε τροπολογία υπέρ 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η τροπολογία 14 καταπίπτει, διότι εγκρίθηκε η συμβαστική υπερθμό 1, η τροπολογία υπερθμό 15 σε δύο τμήματα, επί του πρώτου τμήματος ψηφιπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Ψηφίζαμε τα δύο τμήματα. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Bon, c'est la même chose. Hein. Αμανμό νούμερο 6. Τροπολογία 16. Και εδώ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας πάνω 16 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε. Άρχιτη ψηφοφορία πέρας αυτής. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται 12 ψήφοι υπέρ, 11 κατά. Τροπολογία υπέρ 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπέρ 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 19, 20, 21 και 22 καταπίπτουν, διότι οι τροπολογίες 1 και 2 εγκρίθηκαν. Τροπολογία υπαριθμών 23, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περιθμόν 24. Υπάρχει προφορική τροπολογία του κυρίου Ashworth, ψήφι Κατά. Θα επαληθεύσουμε. Άρχιε ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε 17 ψήφοι υπέρ, 7 κατά. Τροπολογία υπερθυμών 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία υπερθυμών 26. Καταπίπτει επειδή τροπολογία υπερθυμών 2 συμβαστική ενεκτήθηκε. Υπερθυμών 27 τώρα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται η τροπολογία υπαριθμών 30. Υπερ... Υπαριθμών ε, 29-30 τώρα. Ψήφι υπέρ. Ψήφι υπέρ της 30. Ψήφι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά αποχές. Η 31 κατα... έχει καταπέσει. Η 32 επίσης, η 33 επίσης. Συμβαστική τροπολογία υπερθυμών 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική 3 έγινε δεκτή. Τροπολογία υπερθυμών 43. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 47 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία υπερθμών 48. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές το πρώτο τμήμα έγινε δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ σε, ε, συγγνώμη, σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Έγινε δεκτή. Δεν είχαν σηκωθεί όλα τα χέρια. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Προπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε. Άρχιτη ψηφοφορία επί της 55. Πέρασε. Εγκρίθηκε 14 ψήφοι έναντι 9. Τροπολογία συμβαστική 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το υπολογείο υπερθύμων 61. Ψήφι υπέρ, 61, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τώρα επί του συνόλου του κειμένου, όπως έχει τροποποιηθεί, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχισε η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 20 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Σε χαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Νι Ριάντα. Πρώτη συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται δύο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται τρία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται τέσσερα υπέρ κατά, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέντε. Με προφορική του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο Συμβιβαστική δύο υπέρ. Κατά. Δεν σηκώσατε όμως όλοι τα χέρια σας. Θα κάνουμε ονομαστική για τη συμβιβαστική 2. Ψηφίζουμε. Τέλος. Μπορείτε να σηκώνετε τα χέρια σας, σας παρακαλώ. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 με προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 και 11 καταπίπτουν. Συμβιβαστική 4 υπέρ. με ξεχωριστή δεν αντιτίθεται κανείς. Το πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα δεν εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Η κυρία Νηριάντα. Δεν ε, θέλω βεβαίως να καθυστερήσω παραπάνω, αλλά να πω ότι έγινε λάθος στην μετάφραση στην τροπολογία 18. Η αρχική υπευλήθη στα γαλλικά, μεταφράστηκε κατόπιν αγγλικά και ουσιαστικά πήραμε αυτή τη διατύπωση της 18, 19 και 20 για τη συμβιβαστική. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε εδώ την 18. Ουσιαστικά πρόκειται για μόνιμες και όχι αορίστου χρόνου ε, συμβάσεις. Πρόκειται για τροπολογία προφορική που υποβάλλω, δηλαδή μπορεί να σημαίνει το ίδιο στα αγγλικά, αλλά θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι η μετάφραση είναι ακριβής, μόνιμη και όχι αορίστου του χρόνου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνείτε όλοι, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη διευκρίνηση. Ψηφίζαμε το πρώτο τμήμα αυτής της συμβεβαστικής τροπολογίας ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές. Το πρώτο εγκρίνεται λοιπόν. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές και το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 22 εγκρίνεται. 23 και 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται και οι δύο. 25 καταπίπτει. Τη λογική σκέψη. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Έγινε κάποιο λάθος. Επειδή καταπίπτει το δεύτερο τμήμα της τελευταίας τροπολογίας που ψηφίσαμε, θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την 18. Ποιος είναι υπέρ της 18. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Όχι 19. Δεν ψηφίζουμε τη 19. Διότι ενσωματώθηκε στο πρώτο τμήμα της τροπολογίας που ψηφίσαμε. Περνάμε στην τροπολογία 26. Υπέρ της 26. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για τη 30. Τέλος. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. 9 κατά. 31. Καταπίπτει. 32 το ίδιο. 33. Ποιος είναι υπέρ του 33. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 22 υπέρ 2 κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια.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 Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 καταπίπτει. 17 υπέρ. Υπέρ της 17. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18. Α, όχι, να ελέγξουμε. Κύριε Φερνάντες, να ελέγξουμε τη 17. Ψηφίζουμε λοιπόν τη 17. Τέλος. εγκρίνεται 13 υπέρ 10 κατά. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Καταπίπτει. Ψηφίζουμε λοιπόν μόνο το δεύτερο τμήμα. Το πρώτο καταπίπτει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το, τε, το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω να ψηφίζετε όλοι. Θα ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Ελέγχουμε όμως, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, 8 κατά. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του κειμένου ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Τέλος. Εγκρίνεται. 21 υπέρ, 4 κατά, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα περνάμε στην έκθεση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 κατά ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας για την 7. Τέλος. Απορρίπτεται. Οκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εννιά υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Το πρώτο τμήμα. Κατά. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και το δεύτερο. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται το κείμενο 17 υπέρ. 8 κατά. Μία αποχή. Συγχαρητήρια. Δεν θα συγχαρώ τον εισηγητή. Ο κύριος Φερνάνδης είναι ο εισηγητής της επόμενης έκθεσης. Πρόκειται για τις μεταφορές. Πρόκειται για τον προπολογισμό του 16. Πρόκειται για τις μεταφορές πιστώσεων 6 και 7 που απορρέουν ως συνέπεια από τα όσα ψηφίσαμε τώρα για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Μιλούμε για 5 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για χρήματα από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κονδύλια δηλαδή για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Αυτά για το 04-05. Για το 07 επίσης πρόκειται για χρήματα από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αρχικά ήταν το 40-43. Πηγαίνουν και αυτά στο 04-01-04, δηλαδή για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Και εγώ προτείνω και οι δύο αιτήσει για μεταφορές πιστώσεων να ψηφιστούν. Νομίζω ότι κοιτώντα και το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, σας κάνω το αίτημα να ψηφίσουμε για τα δύο κείμενα μαζί. Αρχίζει η ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Τέλο. κλου. Τέλος. Εγκρίνεται το κείμενο. 20 4 κατά. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Νίλ Στόρβαλ, ο οποίος είναι εδώ στη θέση του εισηγητή του κ. Ντεπρέ. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Στόρβαλτς. Πρώτα είναι μία μεταφορά για την Επιτροπή Περιφερειών για το 15.933. 5,4 λέει, αλλά χωρίς να διευκρινίζει τι πράγμα είναι και επίσης για το δικαστήριο, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή μήπως προτιμάτε να τα σχολιάσω ξεχωριστά τις δύο μεταφορές πιστώσεων. Όχι, όλα μαζί. Ο Πρόεδρος, προτείνω να εξετάσουμε τις προτάσεις αυτές ανά όργανο, αναθεσμικό όργανο και να αρχίσουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτοί χρειάζονται για την 4-5-4-0-0-0 που να χωριστεί ανάμεσα στις 2.100 ένα κονδύλιο δηλαδή 400.000 για να αυξήσουν την ικανότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους και 25.000 ευρώ επίσης για την αναβάθμιση άλλων εξοπλισμών. Έχει γίνει πρόοδος τις, ε, τους τελευταίους μήνες, δηλαδή είναι πλέον αποδοτική η υπηρεσία μετάφρασης και γίνεται και συνεργασία διασθεσμικά ή διοργανικά. Θα τους επιτρέψει να κάνουν σημαντικές εξοικονομήσεις. Σύμφωνα με το άνθρωπο 100. Εντάξει, αν δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται αυτές οι μεταφορές χωρίς να χρειαστεί ψηφοφορία. Βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Oui, madame, vous avez Έχετε το λόγο. Εγώ θα ήθελα να ψηφίσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Μία ψήφος κατά. Και τώρα περνάμε στο άλλο θεσμικό όργανο, ο κύριος Τόρβαλς. Για τέσσερις θέσεις συνεργατών, AST δηλαδή, για να μπορέσουν να προσλάβουν νέα μέλη προσωπικού για ε, υπηρεσίες γραμματείας. Το οργανόγραμμα πρέπει δηλαδή να προσαρμοστεί και χρειάζεται να μετατραπούν ορισμένες θέσεις AST σε AST SSE. Και φαίνεται πως θα προκύψουν εξοικονομήσει τη τάξη των 15.000 ευρώ για τον προπολογισμό τη Επιτροπή Περιφερειών του 2016. και ένα ποσό της τάξης των 35.000 για τον προϋπολογισμό του 2017. Έχετε ερωτήσεις ή κάποια αμφιβολία. Άρα, υποθέτω ότι και εδώ θα θέλετε να γίνει ψηφοφορία. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία με νομιστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η μεταφορά πιστώσεως με 20 ψήφους υπέρ, 3 κατά. Θα έρθουμε τώρα στην πολιτική ακινήτων. Αναζητώ με το βλέμμα την εισηγήτρια. Φαίνεται πως η Χολμάιρ δεν είναι ε, ακόμη παρούσα, ίσως όμως έχουμε προχωρήσει ταχύτερα εμείς. Est-ce ο συντονιστής... Όχι, είναι διακοφατικά ο κύριος Φερνάντε. Προτείνω τότε να διακόψουμε για λίγο τις εργασίες μας, αφού δεν έχουμε και άλλο ε, θέμα να ψηφισουμε Sinon, je reporterai ce vote à demain matin. Αλλιώς να αναβάλουμε την ψηφοφορία για αύριο το πρωί, λέει ο Πρόεδρος. Monsieur le coordinateur, quelle est votre observation? Εσείς συντονιστά, ε, τι θα θέλατε να παρατηρήσετε. Αφού δεν είναι παρούσα η εισηγήτρια και δεν είναι δυνατόν να την βρούμε στο τηλέφωνο, ας ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Να ανακοινώσουμε την ώρα της ψηφοφορίας, ώστε να μπορούν όλοι να είναι ακριβείς, 10 το πρωί, αύριο 10. Αύριο λοιπόν στις 10 θα αρχίσει η ψηφοφορία. Δεν έχετε ενστάσεις. Άρα θα ψηφίσουμε περί της πολιτικής ακινήτων αύριο το πρωί στις 10. Και έχω κάθε εμπιστοσύνη στην κυρία Χολμάιρ θα είναι παρούσα αύριο το πρωί στις 10. Άλλα θέματα. Όχι. Διακόπτεται τη συνεδρία μέχρι αύριο το πρωί στις 10.